Ξέρουμε ότι υπάρχει από την κατάσταση αυτή στις Ελληνικέ χώρες ο κίνδυνος εισρωή νέων προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ε, θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε ε, υπόψη για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μελλοντικά προβλήματα. Ευχαριστώ και εδώ κλείνω ο κατάλογο των ομιλητών από τις πολιτικέ ομάδε. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ μια αντιπροσωπεία από τη Βουλή της Βραζιλίας, η επενδυσία του Κάλλος Αλβέρτο Λαρέα, που βρίσκονται στα θεωρείο. Παρακολουθούν την συνάντηση Κοινοβουλίων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας, που είναι ε, ένα βήμα διαλόγου μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Εθνικού Κογκρέσου της Βραζιλίας. Αν είναι δυνατόν αυτές οι αφήσει ε, να αφαιρεθούν, παρακαλώ.

Um, Ζητώ συγγνώμη για το συμβάν αυτό, για την προσωπία παρήσατε στην πρώτη δεκοινοβουλευτική συνεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βάσης, ο κύριος Μπρόκ. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να δούμε τι γίνεται. Ποιοι βουλευτές είναι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για αυτό το συμβάν. Αν έχετε πληροφορίες, οποιοδήποτε έχει πληροφορίες, λέει ο Πρόεδρος, θα μπορούσε να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρει αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα πόστερ θα ε, ήθελε ίσως να επικοινωνήσει με το γραφείο του Προέδρου. Εγώ πάντως θα συνεχίσω, λέει ο Πρόεδρος. Διευθυντικός διάλογος ανάμεσα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του, Ευρω... και του Βραζιλιάνικου Κογκρέσου μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας και επίσης ε, υπάρχει συζήτηση για την συνεργασία με το Mercosur. Καλώ ορίσατε λοιπόν. And the first στη συζήτησή μα, ο κ. Κασουλίδης.